I hope that everybody has kissed everybody. Λοιπόν, ελπίζω να τελειώσανε οι ασπασμοί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, τους φιλήσατε όλους. Πάμε τώρα. Έχουμε και επεξηγήσεις ψήφου. Mr. Ο κύριος Μαμίκινς. Dear colleagues, dear colleagues, we already... Οι ε, συνάδελφοι, έχουμε περάσει επεξηγήσεις. Παρακαλώ πρέπει να ακούσουμε τους συναδέλφους μας που έχουν επεξηγήσει ψήφου να κάνουν. Λοιπόν, έχουμε τη σύσταση της κυρίας Καλνιέτε. Συμφωνία πλαίσιο ξενολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ. Κύριε Μαμίκινς, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπήρου μας έδειξε ότι πρέπει να κάνουμε διάφορες αλλαγές σε διάφορες συμφωνίες που έχουμε με άλλες χώρες για να καλύψουμε τη διεύρυνση. Ε,